για εξωτερικά θέματα για την κατάσταση στην Αιθιοπία. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο εκ μέρους της Αντιπροέδρου στον Επίτροπο κύριο Στυγιαννίδη έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι αυτό το επόμενο ζήτημα ε, εξ της ε, Αντιπροέδρου, κυρία Μογκερίνη, θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας την κατάσταση στην Αιθιοπία τέσσερις μέρες προτού διεξαχθούν οι εκλογές. Είναι σημαντικό να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτήν την τόσο σημαντική χώρα. Ας αρχίσω με αυτά που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει να αναγνωριστεί ενεργός ρόλος και οι περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες της ε, Αιθιοπίας σε σχέση με τις προσπάθειες που κάνει η Αιθιοπία και στο, στα πλαίσια του ΆΙΚΑΤ στο Νότιο Σουδάν και ε, συμμετέχει ε, σημαντικά στην επιχείρηση της Αφρικανικής Ένωσης για τη Σομαλία. η καταπολέμηση της Al-Shabaab με αρκετά μεγάλη επιτυχία μπορεί να αποδοθεί εν μέρη στις προσπάθειες της Αιθιοπίας και αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικός εταίρος είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Έχουμε κοινά συμφέροντα και παρεμφερείς θέσεις για μια σειρά από παγκοσμίων διαστάσεων ζητήματα. Ε, Παραδείγματο χάρη μετανάστευση και εκτοπισμένου πληθυσμού ε, είναι βασική ε, αρχή, χώρα προέλευση, διέλευση αλλά και προορισμού. Η Αιθιοπία επίση πάνω από 680.000 πρόσφυγες είναι σε καταβλισμούς στην Αιθιοπία με όλες τις στις ε, δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται. Εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία Χαρτούμ. Ε, στη Λιβύη ε, η πρόσφατη δολοφονία των χριστιανών έθεσαν το ζήτημα της τρομοκρατίας αλλά και της μετανάστευσης στο προσκήνιο και η κυβέρνηση εξέφρασε ένα ενδιαφέρον για την διεύρυνση της συνεργασίας για αυτά τα ζητήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις κλιματικές αλλαγές, η πολιτική της Αιθιοπίας σε παγκόσμια συζητήσεις ευθυγραμμίζεται με τη δική μας. Έχουμε την πρόθεση να προσυπογράψουμε τη δήλωση της Λίμα για τη συνεργασία με την Αιθιοπία όπως έχουν ήδη πράξει ε, διάφορα κράτη-μέλη. Ως προς την οικονομική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας, θεωρείται η Αιθιοπία από πολλές πλευρές ε, ως ε, μια μεγάλη επιτυχία για την Αφρικανική Ήπειρο. Η βοήθεια που παρέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της στην Αιθιοπία αποφέρουν τους καρπούς τους για την υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας αλλά καθώς και για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής πρόοδου. Βάσει εκτιμήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Οικονομική Ανάπτυξη για το τρέχον έτος 2015 ε, φτάνουμε στο, ε, ε, από το 7,5% έως το 8,5% σε αναπτυξιακό ρυθμό. Είναι μάλλον εντυπωσιακό για αυτή την περιοχή. Επιπροσθέτως, σε βάση Τελευταία έκθεση Παγκόσμια Τράπεζα η ε, φτώχεια στην Αιθιοπία μειώθηκε κατά ε, το 1 τρίτο από το 2000 έως το 2011. Αξιομνημόνευτα επιτεύγματα και πολύ χαίρομαι που συμβάλλουμε και εμείς ε, στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Ξέρουμε όμως ότι αυτό το νόμισμα έχει και άλλη μία όψη, όπως σε πολλές καταστάσεις που δημιουργούνται μετά από έναπλες σειράξεις, η δημοκρατική μετάβαση στην Αιθιοπία διανύει μια δύσκολη περίοδο και δεν εξελίσσεται ομαλά πάντοτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση του ότι το πολιτικό περιβάλλον δεν είναι τέτοιο ώστε ε, να υπάρχει αξιοπιστία, διαφάνεια και αποφύγη αποκλεισμών στην εκλογική διαδικασία. Έχουμε εκφράσει αυτή την ανησυχία μας στις επαφές που είχαμε με την κυβέρνηση βάσει του άρθρου 8, δηλαδή για τον πολιτικό διάλογο και τις διμερείς επαφές, ακόμη και σε ύπατο επίπεδο. Επανειλημμένα έχουμε τονίσει την ανάγκη που υπάρχει να υπάρξει ουσιαστικό πολιτικό διάλογο και με την αντιπολίτευση, ούτω ώστε να γίνεται πλήρω σεβαστή η ελευθερία του συνέχεια της έκφραση και της ελευθεροτυπία, όπως ε, προβλέπει εξάλλου και το Σύνταγμα τη Αιθιοπία. Η γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι πως ε, η πρωταρχική του ανησυχία είναι η σταθερότητα, η ασφάλεια για το λαό της χώρας και ισχυρίζονται πως δεν μπορούν να επιτρέψουν αποσταθεροποίηση της χώρας η οποία ε, θα θέσει εν κινδύνο την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε σε όλα, παρόλα αυτά ε, συνεχίζεται ένας ανοιχτός διάλογος για αυτά τα ζητήματα και ενίοτε έχει και επικοδομητικά αποτελέσματα. Φερρυπίν, συζητούμε τη δυνατότητα συνεργασίας για την βελτίωση της ποιότητας των κρατικών και ιδιωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ως αποτέλεσμα ενός πρόσφατου ε, διαλόγου δυνάμει του άρθρου 8 για τα ΜΜΕ. Ως προς τις εκλογές, η παρακολούθηση της πρόοδου και η εφαρμογή των συστάσεων προηγουμένων αποστολών ε, εκλογικών διαδικασιών δεν ε, έχει ε, συμβεί και στις εκθέσεις του 2005 και ε, αυτό που μας προσέφερε η Αιθιοπία είναι μια απόρριψη και δεν μας απίθυνε καν πρόσκληση για τις εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή και άρα δεν θα στείλουμε ε, αποστολή παρατηρήσεις των εκλογών. Επίσης, αποφασίσαμε έτσι να μην χρηματοδοτήσουμε ε, το, ε, ε, την εκλογική διαδικασία. Η κατάσταση των δημοσιογράφων ε, και άλλων ε, ιδιωτών, bloggers κτλ. είναι πηγή ανησυχίας, έχουν φυλακιστεί διότι εξέφρασαν δημοσίως τις απόψεις τους. Επίσης, ο χώρος που είχαν ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εφημερίδες, παραδείγματος χάρη και στην τηλεόραση, περιορίστηκε ε, κατά την προεκλογική διαδικασία που άρχισε το 2014 ε, σε συνεργασία με την επιτόπου αποστολή μας στην Αντισαμπέμπα παρακολουθούμε στενά αυτά που συμβαίνουν και τις δίκες συζητούμε αυτά τα ζητήματα με τις ε, αρχές ε, καθώς και τη χρήση με την πολιτική για τους αντιφρονούντες ε, που υπάρχουν ισχυρισμοί για τρομοκρατικές ενέργειες γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι η θέση μας η εταιρική μας σχέση με την Αιθιοπία για διεθνή ζητήματα δεν σημαίνει ότι παραμένουμε αδιάφοροι στις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο πληθυσμός στην Αιθιοπία. Ε, όπως συζητήσαμε και στον Ιανουάριο στην Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, το 2015 καθώς και το Σεπτέμβριο του 2014 προκύπτει ότι έχουν γίνει δύο δηλώσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Αιθιοπία από πλευράς Επιτροπής και σίγουρα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε δημοσίως όταν χρειάζεται. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για τις σχέσεις μας με την Αιθιοπία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed, ε, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα από πλευρά του ΕΛΚΑ ο κύριος ε, Ντάβο Ρίβο Στήρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Αιθιοπία έχει 94 εκατομμύρια κατοίκου είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες τη Αφρικής και είναι χώρα κλειδί για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Υπήρου. Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντική και για την ευρωπαϊκή μας ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό το γεγονό ότι αναφέρεται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς και ανησυχούμε ιδιαίτερα για τους διάφορους περιορισμούς ε, των δημοκρατικών ελευθεριών ε, στην Αιθιοπία και την ε, κράτηση δημοσιογράφων, blogger και άλλων. Στην Αιθιοπία διαπιστώνουμε, όπως και σε άλλες αφρικανικές χώρες, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της διαχείρισης της ε, πολιτικής της μείωσης της ένδυας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό και ακριβώ θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι εκλογές ε, να είναι ελεύθερες και πριν από τις εκλογές οι αντιφρονούντες ε, να ε, αποφυλακιστούν. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα την ανάπτυξη της χώρας βοήθειά μα τώρα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε ω εταίροι στην περιοχή αυτό. Και, ε, και γιατί αυτό. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Αιθιοπία να συνεχίσει ε, την επικοδομητική περιφερειακή συνεργασία. Παρά το γεγονό ότι η χώρα αυτή είναι πάρα πολύ φτωχή και έχει πάνω από 680.000 πρόσφυγε στη χώρα τη, είναι πολύ σημαντικό για την Αιθιοπία να συνεχίσει να δίνει μάχη κατά της τρομοκρατίας. Ε, και επειδή ακριβώς θέλουμε η τρομοκρατία να είναι ισχυρό, η Αιθιοπία συγγνώμη, να είναι ισχυρός εταίρος, θα πρέπει να ενισχύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εφαρμογή του κράτους δικαίου και ελπίζουμε η κυβέρνηση να ξεκινήσει ένα αξιόπιστο διάλογο με την αντιπολίτευση, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Κιέγκε. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Αιθιοπία είναι σημαντικός παράγων για, την ειρήνη στο κέρας της Αφρικής, για τη Σομαλία, την Ερυθρέα, τον Νότιο Σουδάνα. Αλλά για να μπορέσει να διαδραματίσει αυτό το διεθρή ρόλο που της αντιστοιχεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ειρήνη και στο εσωτερικό της χώρας. Δεν μπορεί να υπάρξει βοήθεια προς την ανάπτυξη χωρίς να ξεκινήσει μια διαδικασία εκδημοκρατισμού της χώρας. Η Αιθιοπία ε, θα ψηφίσει την Κυριακή όπως ακούσαμε. Ε, η, το αποτέλεσμα όμως των εκλογών αυτών το γνωρίζουμε ήδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να μην στείλει παρατηρητές για αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε οι κύριοι χορηγοί ε, αυτής της χώρας και επομένως έχουμε καθήκον και ευθύνη να επαγρυπνούμε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαφορετικότητα, καθώς επίσης και την καλή διακυβέρνηση δίνοντας κίνητρα για την διαδικασία του εκδημοκρατισμού. Είναι πάμπολες οι καταχρήσεις που γίνονται στη χώρα αυτή. Υπάρχουν ε, νέοι φοιτητές ε, σπουδαστές, διδάσκοντες ε, και οι οποίοι έχουν συλληφθεί από την κυβέρνηση της Αιθιοπίας και αυτό τα στοιχεία μας έδωσε η Ένωση για τα Δικαιώματα των ε, Ανθρώπων ε, στο κέρας της Αφρικής. Είχαμε 20 τραυματίες μόνο τον Απρίλιο σε μια χώρα όπου ε, συλλαμβάνονται ε, blogger, όπως ο blogger ο οποίος συνελήφθη από το blog ε, Ζώνη 9, ο οποίος βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο στη φυλακή. Κάθε μέρα υπάρχει εκφοβισμό δημοσιογράφων και blogger. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο δεν αποτελεί ένδειξη. Αυτό το είδανε ο Γιώχαν Πέρσον και ο Μάρτιν Βίτζερ, Σουηδοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν το 2011 και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από 14 μήνε φυλάκισης. Η Ευθεοπία βιώνει αυτή τη στιγμή μια οικονομική ανάπτυξη. Επομένω, ε, πρέπει και το καθεστώ να οδηγηθεί προ μια πιο ισότιμη κοινωνία που θα σέβεται τα δικαιώματα του ατόμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο... Από πλευρά του ΙΣΙΑ, ο κύριος Πετρόφσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, ε, σε λίγο θα γίνουν ε, εκλογές στην Αιθιοπία. Και ναι, παρατηρούμε εδώ και πολύ καιρό παραβιάσει και περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ελευθερία έκφραση. Και ναι, μεν όπω είπε και ο Επίτροπο, ε, έχουμε παρατηρήσει τέτοιου περιορισμού, εξακολουθούμε να του στέλνουμε αναπτυξιακή βοήθεια και άλλε χρηματοδοτήσει από τον Ιδρυσιακό Ταμείο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τουλάχιστον ένα αποτελεσματικό έλεγχο αυτών των δαπανών, διότι ε, έχουμε προβλήματα με του εξωτερικού παρατηρητέ ε, των εκλογών. Ε, είναι σημαντική για μα η Αιθιοπία, κυρίω για λόγου μετανάστευση πρόσφατα, όπως ξέρετε, οι Ισλαμιστές στη Λιβύη δολοφόνησαν κτηνοδός 30 χριστιανού ε, στη Λιβύη λοιπόν και αυτό δημιούργησε αναταραχή στην Αιθιοπία. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε μια αποστολή παρατήρηση παρά το ότι δεν έχουμε προσκληθεί. Διότι αυτή η κοινωνική αναταραχή θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη χώρα που είναι μία από τις πιο πολυπληθείς χώρες της Αφρικής και από όπου έρχονται πολλοί ε, παράνομοι μετανάστες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Για ε, για την προηγούμενη επιτροπή ο Επίτροπος κύριος Μισελ. Ε, ναι, μόλις ε, επέστρεψε από μια αποστολή στην Αντίς όπου συζήτησαμε τον Πρωθυπουργό για τις προσεχείς εκλογές και την κατάσταση στη χώρα και την περιοχή ευρύτερα. Και η εντύπωση που έχω, η άποψη που έχω για τον Άιλε Μαράμ Ντεζελέγκ είναι ότι είναι ένας Πρωθυπουργός που είναι πάνω από τις διαμάχες. Έχει το προσόν ότι δεν τον αφορούν οι εθνοτικές αλλά και θρησκευτικέ ε, διαμάχες. Είναι μουσουλμάνος, ενώ σε λαού είναι χριστιανός και παρόλα αυτά είχαν πολύ καλές σχέσεις. Αυτό λοιπόν είναι σίγουρα πλεονέκτημα. Έχει περίπου 5.400 χιλιόμετρα σύνορα η Αιθιοπία και αυτό σημαίνει ότι εξαρτάται πολύ από την ε, έλλειψη σταθερότητα ε, στι γειτονικέ χώρε. Και ξέρετε ότι επίση είναι στόχο των γειτονικών Ισλαμιστικών πιέσεων και έχει αποδεχθεί από το 2014 οι δυνάμεις της να παρεύουν στη Σομαλία στα πλαίσια της Αφρικανικής Ειρηνευτικής Δύναμης. Είναι λοιπόν ουσιώδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει έναν έντονο πολιτικό διάλογο με τη χώρα αυτή γιατί είναι χώρα κλειδί για την περιοχή. Υπενθυμίζω ότι έχει ε, πάνω από 90 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι γίγας στο κέρας της Αφρικής και παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθερότητά του. Οι Ηνωμένε Πολιτείε το έχουν κατανοήσει εδώ και πολύ καιρό και στηρίζουν τη χώρα. Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε την Αιθιοπία για να παίξει ηγετικό ρόλο κατά της τρομοκρατίας στην περιοχή. Η χώρα αυτή έχει αναπτυχθεί, έχει βελτιωθεί από την ε, οραματική προσέγγιση του Μέλε Σελαγουή, του προκατόχου του σημερινού Πρωθυπουργού, που φαίνεται ότι αποτελεί συνέχεια και θέτει την υπευθυνότητα και την νεότητα στο κέντρο των προσπαθειών του. Αλλά βεβαίω ε, πρέπει πολλά να κάνουμε ακόμη για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα μελανό σημείο. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο ενό ε, προνομιακού διαλόγου με αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ η Λίδια Σένδρα Ροντρίγκες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να λέμε ότι η Αιθιοπία είναι μοντέλο εκρίζωσης της φτώχειας της περιοχής όταν ε, αναφερόμαστε σε μια χώρα που έδωσε στα χέρια ξένων επιχειρήσεων πάνω από 100.000 ε, στρέμματα. Ε, όταν αναφερόμαστε σε μια κυβέρνηση που προχωράει ε, προγράμματα τα οποία κατασκευάστηκαν από μια Ιταλική πολυεθνική και κάνει τεράστιες εκθέσεις όπως το κουράθ που απειλούν τον ποταμό Όμο που είναι ε, ο ποταμός από τον οποίο ζουν ε, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που ζουν από το ποτάμι και από την κοντινή ε, λίμνη και δεν τους επιτρέπουν να αντισταθούν σε όλες αυτές τις κατασκευές. Αυτό θα δημιουργήσει περισσότερη πείνα, περισσότερη ένδυα σε μια χώρα στην οποία ήδη το 80% ζει με κάτω από 2 δολάρια την ημέρα. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μοντέλο για τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όχι για τα συμφέροντα των ανθρώπων που ζουν στη χώρα χώρα αυτή. Θα ήθελα σας παρακαλώ να διαβιβάσετε στην κυρία Μογκερίνη εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδος ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τόλο σε αυτή την ε, δυτική ε, πλεονεξία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταπολεμήσουμε αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ εκ μέλους των Πρασίνων. Ο Γιώργη Σεμπάστια, για 1,5 λεπτό. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τελώ υποσύγχυση. Μου περιγράψατε μια ενθεωπία την οποία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζω. Όλοι ξέρουν ότι οι εκλογέ τη Αιθιοπία είναι μια φάρσα. Είναι μια από τι χώρε η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρατηρητέ των εκλογών που εστάλησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν δικαίωμα πρόσβαση. Σουηδοί δημοσιογράφοι είναι στη φυλακή απλώ και μόνο γιατί μπήκαν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ε, ανα, υπάρχουν ε, συνεχείς καταγγελίες για τη δίωξη των ε, μελών της αντιπολίτευσης, των δημοσιογράφων που καταγγέλουν την κυβέρνηση, πολιτικών ομάδων, τον ομο, Όμο, τον Ογκαλέν, τον Σιράμα και δεν επιτρέπεται να μπουν παρατηρητές και δημοσιογράφοι στην περιοχή του Ογκαλέν, όπου ε, αναφέρεται ότι 30% των γυναικών βιάστηκαν από κυβερνητικούς παράγοντες μάλιστα. Ε, και ε, θα ήθελα να ζητήσουμε ε, πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση τη Αιθιοπία. Θα πρέπει να υπάρξει μια αποστολή η οποία θα διερευνήσει τα θέματα τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι διώξει και του βασανισμού. Ε, ο λαός της Αιθιοπίας δεν θα πρέπει να υποφέρει ε, από μια κυβέρνηση την οποία ανέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κανένα τμήμα της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα δίνεται για όλη αυτή την καταπίεση. Έχουμε πολύ σημαντική ευθύνη για το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν. Θα είμαστε συνένοχοι και θεωρώ ότι ήγηκε και η ώρα να τράψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του EFTD, ο James Carver, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν ανησυχίε εδώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αιθιοπία. Και είναι σωστό ότι θα πρέπει να την ενθαρρύνουμε να σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών τη. Αλλά θα ήταν ανόητο να θεωρήσουμε ότι εμεί τα ξέρουμε όλα. Α πάρουμε το θέμα, για παράδειγμα, που ε, πάρουμε το θέμα ότι πολλές φορές μετακινούνται ε, πολλοί πληθυσμοί από το χωριό τους για να ε, γίνει εμπορική εκμετάλλευση. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε στο καθρέφτη πριν ε, αποφασίσουμε εάν υποστηρίξει η πολιτική, υποστηρίζει αυτή η πολιτική αυτές τις ενέργειες. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Αιθιοπία έχει υποδεχθεί 650.000 πρόσφυγες πληθυσμούς από το Νότιο Σουδάν, την Ερυθρέα και τη Σομαλία. Η Ιθιοπία έχει καλές σχέσεις με τη Δύση. Είναι ουσιώδες λοιπόν αυτή η ισχυρή δύναμη σε αυτή την περιοχή του κόσμου που έχει τόσα προβλήματα να μπορέσει να συνεχίσει να αναπτύσσει την οικονομία της για να προωθηθεί η σταθερότητα στην περιοχή μαζί με το γείτονά της την Σομάλιλεν που θέλει την διεθνή αναγνώριση που όντως της αξίζει αντί να αντιδρούμε σπασμωδικά και για να αντιμετωπίσουμε την ε, περαιτέρω μεταναστευτική ροή θα πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει καταστροφικό ρόλο στην περιοχή. Όπως ξέρετε, ο καφές είναι το 28% των εξαγωγών και αντιμετωπίζει ε, δασμούς του 9%. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε την ε, χώρα, πρέπει να σταματήσει αυτός ο προστατευτισμός και να ε, βοηθήσουμε να ξάγει καφέ αυτή η χώρα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Μαρή Κριστίνα Γλωτσού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν οι ψηφοφόροι της ε, Αιθιοπίας, αλλά πολύ πιθανό είναι ότι θα συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός ο σημερινός πρωθυπουργός. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ένωσης να στηρίξουν την κυβέρνηση της Αιθιοπίας. Είναι μια σπάνια νησίδα ανάπτυξης και σταθερότητας στην Ανατολική Αφρική. Διότι μέχρι στιγμής είμαστε μεγάλοι απόντες. Αφήνουμε την Κίνα ε, να δρά ανεξέλεγκτα στην Αιθιοπία. Πρέπει να βοηθήσουμε την ανάπτυξη. Πρέπει να εγκατασταθούν ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη χώρα και πρέπει να συνεργαστούμε πιο ενεργά και μάλιστα στρατιωτικά με την Αιθιοπία για την καταπολέμηση του ακραίου Ισλαμισμού και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των συνόρων της χώρας. Και ως αντάλλαγμα πρέπει να ζητήσουμε από την Αθιοπία περισσότερη αποτελεσματικότητα στην ε, καταπολέμηση της ε, παράνομης μετανάστευσης ιδιαίτερα μέσω της Λιβύης που θέτει εν κινδύνο τους μετανάστες που ε, εκτός από τον πνιγμό από τον οποίο κινδυνεύουν στην Μεσόγειο μπορεί να δολοφονηθούν και από το Ισλαμικό κράτος στις χώρες διέλευσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριος Βέντα για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 24 Μαΐου θα γίνει θα προσέλθουν οι Αιθιώπες στις κάλπες ε, για να ψηφίσουν και υπάρχουν φόβοι ότι δεν γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα και μπορεί να μην είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα των εκλογών λόγω της, της εκλογικής διαδικασίας. Η πολιτική πολυφωνία στη βάση της δημοκρατίας για να γίνουν εκλογές ε, θα πρέπει ε, να είναι μια διαδικασία ανοιχτή και ισότιμη που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους. Γι' αυτό ακριβώ η κυβέρνηση της Αιθιοπίας θα πρέπει να διασφαλίσει μια πολιτική συζήτηση που θα είναι ανοιχτή για όλους και να γίνει σεβαστός εκλογικός νόμος. Η καταπολέμηση της, δημοκρα... της διαφθοράς και η ελευθερία του λόγου είναι δύο θεμελιώδη δικαιώματα προκειμένου να υπάρχουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Αλλά οι αρχές της Αιθιοπίας βίας, ε, ε, διώκουν την αντιπολίτευση και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Μπλόγκερ και δημοσιογράφοι βρέθηκαν στη φυλακή αυθαίρετα. Υπάρχει διάκριση κατά των χριστιανών και παραβίαση των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων. Ε, σεξουαλική καταπίεση επίσης είναι όλα αυτά θέματα τα οποία υπάρχουν και πολλές από αυτές τις διώξεις γίνονται από το στρατό της Αιθιοπίας. Η Συμφωνία του Κοτονού για την ελευθερία της έκφρασης, για την ελευθερία, τα πολιτικά και ε, προσωπικά δικαιώματα τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά. Και υπάρχουν επίση κατηγορίε για βία, για ε, σεξουαλική βία, βιασμού και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταδικάσουμε. Σα ευχαριστούμε για αυτή την τόσο σημαντική παρέμβαση. Και τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Βάδεν Χόλτσερ. Ένα λεπτό μάλλον. Ευχαριστώ. Το κέρας Αφρική για την ασφάλειά μα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η Αιθιοπία είναι κεντρικό στοιχείο. Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας μας δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και γι' αυτό ε, επενείται από πλευράς μας οι εκλογές, οι λεγόμενες εκλογές, φαίνεται ότι εξυπηρετούν τη συνέχιση αυτού του ρόλου. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ασφάλεια δεν σημαίνει ησυχία νεκροταφείου. Η μόνιμη ασφάλεια σημαίνει κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και όλοι να μπορούν να εκφραστούν. Και αυτό που με ανησυχεί εμένα και πολλούς άλλους είναι η κατάσταση των καντέν. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες, εάν δεν επιχειρήσουμε να αλλάξει η κατάσταση, τότε στην ουσία προετοιμάζουμε το έδαφος για τον εξτρεμισμό. Μόνο λόγω αυτής της φαινομενικής ασφάλειας δεν καταπολεμούμε τον εξτρεμισμό στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρο. Και τώρα ο κύριος Καστάλντο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 24 Μαΐου θα γίνουν νέες εκλογές στην Αιθιοπία, τη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής. Θα είναι άλλη μια φάρσα και δυστυχία στις εκλογές, διότι οι δημοσκοπήσεις ε, θα μας πούνε αν το κόμμα το οποίο έχει τη, ε, τα ενία της κυβέρνησης, το PRDF, θα έχει το 98, το 99 ή το 100% των εδρών. Η χώρα αυτή έχει ρεκόρ ε, συλληφθέντων δημοσιογράφων σε όλη την Ήπειρο. Εγώ προσωπικώς ε, υπήρξα παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές στην Τινησία και στην Αλγερία, στην Αφρική και είδα στα μάτια αυτών των ανθρώπων τι σημαίνει η ελπίδα για μια πραγματική δημοκρατία. Και σας λέω αγαπητοί συνάδελφοι ότι δεν αρκεί μια οικονομική ανάπτυξη διψήφια και κάποιοι στρατιώτες για να ξεχάσουμε τι ακριβώς είναι και πώς παραβιάζεται καθημερινά το κράτος δικαίου και οι πολιτικές ελευθερίες ε, στην Αιθιοπία. Θα πρέπει να το αναρωτηθούμε και εμείς και θα πρέπει να ζητήσουμε και το ίδιο και από την Κίνα που ε, καταλαϊλατεί τη χώρα. Θα πρέπει να επιδείξουμε συνέπεια στις αξίες μας, ε, οποιοδήποτε και να είναι το κόστος. Ευχαριστώ. Τώρα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Αιθιοπία έχει αναδειχθεί σε πάρα πολύ μεγάλη περιφερειακή δύναμη και πόλος σταθερότητα στο τη της Αφρικής. 10,5% αναπτυξιακός ρυθμό για το 2013. Βλέπουμε τους καρπούς μιας ανάπτυξης που ιδρύεται σε μια κατευθυνόμενη οικονομία από ένα ισχυρό και διαρθρωμένο κράτος. Σε μια Αφρικανική υπηρεσία από διάφορους εμφυλίους πολέμους ε, και απόπειρες επραξικοπημάτων ε, είναι μοντέλο η Αιθιοπία για την πολιτική πολιτική σταθερότητα και παρά τη μεγάλη ε, θρησκευτική και εθνοτική επικοινομορφία τη. Ε, οι εκλογέ που θα διεξαχθούν την Κυριακή είναι οι πρώτε ε, από το θάνατο το 2010 του του πρώην Προέδρου Ζενάουι. Δεν θα πρέπει όμω να αποτελέσουν πρόσχημα για οποιαδήποτε ηθικού τύπου παρέμβαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των δυτικών χωρών στι εγχώριε συζητήσει μια ομολογουμένω απολυτεργική κυβέρνηση, η οποία όμως έχει επιτύχει θεαματικά αποτελέσματα για την καταπολέμηση της ένδυας. Ε, οι ταραχές ε, θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε ένα κύκλο αποσταθεροποίησης, τι ε, τις οποίες την έκφαση κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποδίδουν τη δέουσα έμφαση στο οικονομικό δυναμικό της Αιθιοπίας και καλά θα κάναμε να εντατικοποιήσουμε τις οικονομικές νομικές μας σχέσεις με ίσους όρους. Σας ευχαριστούμε. Η Ελέσια Μαρία Μόσκα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε προσπάθεια από πλευρά Αιθιοπία να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση τη φτώχεια, ε, υποστήριξη τη ανάπτυξη και τη ευημερία που αναγνωρίζουμε και επικροτούμε, μπορεί να υπονομευθεί πολύ σοβαρά εάν ταυτόχρονα δεν υπάρχει και μια προσπάθεια προκειμένου να έχουμε μια βιώσιμη δημοκρατική ανάπτυξη. Και δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια ανάπτυξη αν περιορίσουμε την ελευθερία τη έκφραση και ενημέρωση, που είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη και επομένω είναι και μία από τι βασικέ αξίες επί των οποίων έχουμε οικοδομήσει ε, τη συλλογική μας διαβίωση. Γι' αυτό και ακριβώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να σιωπήσουμε για τα όσα συμβαίνουν εν στην Αιθιοπία και ιδίως εν ώψη των επόμενων εκλογών. Η οικονομική κατάσταση δεν μπορεί να κρίνεται ανεξάρτητα και δεν δικαιολογεί καμία δράση καταπίεσης ε, των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καθήκον να μην αφήσει μόνους τους τους πολίτες και τους δημοσιογράφους, γιατί και έτσι θα βοηθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ. Euh, Julie Ward. Η Julie Ward, παρακαλώ για ένα λεπτό. Θα ήθελα να ευχάρε στήσω τον κύριο Βάτιν Χόλτσερ και άλλους συναδέλφους που μίλησαν για αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν φτάνει αυτό το ζήτημα στα mainstream με μέσα μαζική ενημέρωση. Εγώ συνεργάζομαι με οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών στην Αιθιοπία και είναι σημαντικό να αναφέρω ότι για τι φωνέ αντιπολίτευση δεν υπάρχουν ίσοι όροι. Την επόμενη εβδομάδα γίνονται οι εκλογέ χωρί αποστολή παρατήρηση. Υπάρχει καταστολή των δημοσιογράφων και τη κοινωνία των πολιτών που πλευρά τη κυβέρνηση. Ε, διώκονται διάφορε εθνοτικέ διαφορετικές ομάδες ε, μεταξύ των οποίων ε, και παιδιά και ε, η περιοχή ο Οκτουνά έχει πλέον αποκλειστεί από την ίδια την κυβέρνηση. Στο μεταξύ είναι η τέταρτη στη σειρά η Αιθιοπία σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια και 45% του προϋπολογισμού προέρχεται από εξωτερική βοήθεια. Θα πρέπει να γίνει δημόσια δήλωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις ανησυχίες της για την έκβαση των εκλογών πριν τις 24 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό τους, καθώς και την αλληλεγγύη προς το λαό της Αιθιοπίας ε, τα χρήματα της αναπτυξιακής βοήθειας δεν θα πρέπει να ε, ε, χρησιμοποιούνται για παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για καταχρήσεις. Μία πιο ειρηνική Αιθιοπία δεν μπορεί να γίνει με κόστος της έλλειψης υγιούς αντιπολίτευσης νοθευμένων εκλογών και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστούμε. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Κάρβερ. Ναι. Κυρία Ward, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κάρβερ. Επαναλαμβάνω, δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κάρβερ. Παρακαλώ κύριε Κάρβερ. ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Γουόλ που δεχτήκατε το ερώτημά μου. Ενώ όλοι ανησυχούν εδώ πέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ισχυρισμούς ε, παραβίασης, ε, δεν συμφωνείτε ότι η μεγαλύτερη απειλή ε, είναι ο Ισλαμικός φονταμεταλισμός για το κέρας της Αφρικής και δεν συμφωνείτε ότι θα πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα στην Αιθιοπία για τα όσα κάνει για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού σε αυτό το τομέα, χάρη στην οποία έχει μια πολύ καλύτερη προσέγγιση για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών από ότι κάποιοι εξτρεμιστές, ισλαμιστέ φονταμεταλισμού ε, παρακαλώ κύριε Ward. Κοιτάξτε, εγώ συνεργάζομαι και δαπανώ πολύ χρόνο για ε, τη συνεργασία με ε, αυτούς που, τον οποίο η φωνή συνήθως δεν ακούγεται από την φωνή, συγγνώμη, από την κοινωνία των πολιτών. Και οι οργανώσεις ε, με τις οποίες συνεργάζομαι ε, αναφέρουν ε, σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένα βιασμούς γυναικών και κοριτσιών, παραβίαση των δικαιωμάτων από πλευρά της κυβέρνησης. Ναι, εγώ υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και μία από, από τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια είναι ότι δεν υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση στον κόσμο. Τα δύο φύλλα δεν δεν εκπροσωπούνται ισότιμα και αυτό είναι βασικότατο πρόβλημα στην κοινωνία μας. Μα όντως σας απάντησα. Η μεγαλύτερη απειλή, κύριε Κάρβερ, είναι ότι ε, το παιχνίδι, την ισορροπία των δυνάμων την αποφασίζουν οι άντρες. Τώρα η κυρία Αναγκόμες, δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Οι Αιθιοπίες ε, στην Αιθιοπία που έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Μαΐου δεν θα είναι ούτε δίκαιε ούτε ελεύθερες, ούτε δημοκρατικές. Ε, οι συστάσεις ε, των αποστολών παρατηρήσει το 2005 και 2010 δεν έγιναν σεβαστές από την κυβέρνηση. Αυτή, είναι η πραγματική αιτία για την οποία δεν θα υπάρξει φέτος αποστολή παρατήρησης και όχι όπως λέει στην προπαγάνδα του η κυβέρνηση ότι πρόκειται για οικονομικούς λόγους ε, που ε, αιτιολογούν αυτή την απουσία αποστολής. Λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ε, το EPRFD ε, έχει υπονομεύσει ε, τους προσπάθειές τους για να καταχωριστούν ως υποψήφοι και με μέλη της αντιπολίτευσης διώκονται και έχουν συλληφθεί. Ο μοναδικός ηγέτης της αντιπολίτευσης θα μπορέσει να αναμετρηθεί λόγω της παρέμβασης του κράτους. Η πολιτική πολυφωνία και η ελεύθερη έκφραση και η ελευθεροτυπία είναι πολύ πιο περιορισμένη σήμερα σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν πριν από 10 χρόνια. Ποτέ δεν υπήρχαν τόσοι ε, bloggers, τόσοι δημοσιογράφοι που έχουν ε, προφυλακιστεί γιατί κατηγορούνται για ε, τρομοκρατία. Η Αιθιοπία λαμβάνει τη μεγαλύτερη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σύμμαχος κλειδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης για θέματα ασφάλειας στην περιοχή. Αυτό εξηγεί και την επίκαια που δείχνουμε ενώπιον αυτών των βαρύτατων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ε, θέσπισης αυτών των αντιδημοκρατικών νομοθεσιών, ε, κυρίως στην περιοχή του Αγκαβέν ε, και την καταπίεση των μειονοτήτων. Θα πρέπει να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση της Αιδιοπίας να αποφυλακίσει όλους τους αντιφρονούντες συμπεριλαμβανομένου και του Ανταρκάτσιου Τσίγκε που είναι Βρετανός πολίτης και είναι ηγέτης αντιπολίτευσης σε εξορία, ο οποίος είναι φυλακισμένος από τον Ιούλιο του 2014 στην Ιεμένη και έχει απελαθεί από την ε, η Αιθιοπία. Διατηρούνται λοιπόν αυτές οι εντάσεις από την κυβέρνηση και αυτό είναι αντιπαραγωγικό για τα συμφέροντα της Αιθιοπίας και τα δικά μας. Είναι στρατηγική σημασία της Αιθιοπίας στην περιοχή, δεν μπορεί να σιωπούμε. Πρέπει να απαιτούμε αλλαγή ε, καμπή στην πολιτική που ακολουθούμε για την Αιθιοπία, διότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επιρροή και μπορούμε να κάνουμε την διαφορά, κύριε Στυλιανίδη. Σας ευχαριστούμε. Τώρα Περνάμε στην ε, διαδικασία προσέλγησης του Προέδρου. Η κατάσταση στην Αιθιοπία είναι ενισχυτική από διάφορες απόψεις. Την Κυριακή θα γίνουν ε, βουλευτικές εκλογές στην ε, Αιθιοπία. Ο πλουραλισμός είναι απλώς επιφανειακός τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν σοβαρές ε, διώξεις και περιορισμούς. Και οι δημοσιογράφοι έχουν να διαλέξουν μεταξύ της αυτολογοκρισίας και των διώξεων και πολλοί πρέπει να καταλήψουν τη χώρα. Βεβαίως η χώρα είναι κυρίως ε, χριστιανική, αλλά υπάρχουν διώξεις ε, χριστιανών σε αυτή τη χώρα διότι διώκονται από διάφορους ε, μουσουλμάνους εξτρεμιστές που θέλουν να δημιουργήσουν ένα Ισλαμικό κράτος. Βεβαίως ε, το Κοράνι δεν δικαιολογεί αυτές τους τις αξιώσεις αλλά λένε απλώς ότι έχουν τη στήριξη του Θεού. Πρέπει να καταπολεμήσουμε όλες αυτές τις τάσεις. Η Γεωργία βεβαίως είναι πολύ σημαντική για τον πληθυσμό και αυτή διασφαλίζει την επιβίωσή του. Γι' αυτό πρέπει ταχύτατα να σταματήσουν οι δασμοί για τα προϊόντα που εξάγει αυτή η χώρα. Ο κύριος Νικόλα Καπούτο. Γίνονται πολλά ακόμα για την εθνική ποιά. Πρόκειται για μια χώρα του κέρατος της Αφρικής με πολύ σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και έχει άτομα με ε, το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής. Φτάνουν στα 29 χρόνια και υπάρχει και λειψιδρία. Ακόμα και σήμερα οι γυναίκες πρέπει να διανύσουν χιλιόμετρα για να φτάσουν στις ελάχιστες ε, πηγές και πηγάδια και κάθε μέρα ένα άτομο τουλάχιστον ε, σε κάθε πέντε λεπτά πεθαίνει από έλλειψη νερού. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό μετανάστευση γεγονό το οποίο υποχρεώνει ακόμα και μορφωμένου νέου να διαφύγουν από τη χώρα αναζητώντας κάπου αλλού μια καλύτερη ζωή. Η δύσκολη συμβίωση επίση μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων είναι πρόβλημα. Η κυβέρνηση Τις τελευταίες ημέρες παρουσίασε ένα πολύ σημαντικό σχέδιο επενδύσεων για βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά εάν δεν λυθούν ε, πρώτα τα κατεπήγοντα θέματα τα οποία δεν επιτρέπουν στους ε, ανθρώπους να ζουν με ε, αξιοπρεπέ επίπεδο ζωής, δεν αρκούν οι επενδύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει και συνθήκε βιωσιμότητας. Ευχαριστώ. Ο Νότης Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, στις 19 Απριλίου το ίσις δημοσιοποίησε βίντεο με τον αποκεφαλισμό στη Λιβύη 30 χριστιανών από την Αιθιοπία προκειμένου να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό της αιθιοπίας όπου τα δύο τρίτα των εκατό εκατομμυρίων κατοίκων της είναι χριστιανοί. Στόχο των τζιχαντιστών είναι να χρησιμοποιήσουν και στην αιθιοπία τη θρησκεία και τη φτώχεια για να προωθήσουν τα σκοτεινά τους συμφέροντα. όμως σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες και γυναίκες της αιθιοπίας αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους που πλήττεται από τη φτώχεια την ανεργία την πολιτική αστάθεια και τις συλλήψεις αντιφρονούντων. πρέπει λοιπόν να διασφαλιστούν οι όροι διεξαγωγής δημοκρατικών εκλογών η ελευθερία του τύπου και τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης. ανησυχούμε λοιπόν σοβαρά για την κατάσταση της πολυπληθούς αυτής χριστιανικής χώρας και η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής στην οικονομική ανάπτυξη της αιθιοπίας στη λειτουργία του κράτους δικαίου και στην προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων. πρέπει επιτέλους η αιθιοπία να πάψει να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι για τις μεγάλες κινεζικές και ιταλικές πολυεθνικές επιχειρήσεις. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ιβάν Ο κύριος Ιάκοφτσιτς. Παρακαλώ. Βεβαίως ισχύει ότι εδώ μόνο συζητάμε. Η συζήτηση που κάνουμε είναι παρόμοια αυτή που κάναμε για την Τουρκία. Πρέπει να πούμε τι θετικό υπάρχει στην Αιθιοπία, τι θα βοηθήσει την Ευρώπη Κοιτάξτε, η Αιθιοπία είναι ιδιαίτερα πολυπληθής χώρα και είναι παράγον σταθερότητα σε μια ιδιαίτερα ασταθή και ταραγμένη περιοχή. Και αυτό σημαίνει ότι η στήριξή της στηρίζει τα δικά μας συμφέροντα με κάποιο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Αιθιοπία, αλλά συμφωνώ και με αυτό που είπαν διάφορες συναδέλφοι. Πρέπει να καταδικάσουμε τις αντιδημοκρατικές συνέργειες της παρούσας κυβέρνησης. Αλλά σας παρακαλώ όλους, όταν συζητάμε για την Αιθιοπία και την Τουρκία, να χρησιμοποιούμε τα ίδια μέτρα. Γιατί είναι μια χώρα που είναι πολύ σημαντική για μας. Ο Τζαν Μπονάνο, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, δεν ε, άκουσα το όνομά μου, κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα τη συζήτηση και εδώ ανάλογα με το ποιο μιλάει, κάποιο μα λέει ότι η Αιθιοπία είναι μια καταστροφή, κάποιοι άλλοι έχει ΑΕΠ ε, ανάπτυξη στο 10%, μακάρι να έχει 10% ανάπτυξη η Ευρώπη. Κάθε τόσα λεπτά μα λένε πεθαίνει ένα Αιθιόπιο και ο άλλο μα λέει ότι η Αιθιοπία βγαίνει από τη φτώχεια. Συμφωνήστε επιτέλου και μάλλον αντί να μιλάμε για την Αιθιοπία θα έπρεπε να μιλάμε για περισσότερη Ευρώπη, να μιλάμε για του ηλικιωμένου μα, για του νέου μα που είναι άνεργοι και για τη Λιβύη όπου όλοι οι Ευρωπαίοι που συζητούν εδώ, οι υποκριτές, βομβάρδισαν τη Λιβύη και αυτή τη στιγμή έχουμε το έσχος αυτό στην Λιβύη. Έσχος. Καταφτάνουν οι λαθρομετανάστες με τους τρομοκράτες, με τα σκάφη όπως έγινε σήμερα στην Ιταλία και έχουμε μια κυβέρνηση παλιάτσων στην Ιταλία που μας λέει ότι δεν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η Αφρική που βοηθάει η Ευρώπη. Ξυπνήστε. Ε, Ευχαριστώ τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, ο κύριος Φροντζούλικα. Πάντοτε ε, χαιρόμαστε όταν προεδρεύεται η Αιθιοπία είναι ε, πολύ σημαντικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες τις πλευρές, έχει στρατηγική θέση στην περιοχή και ρόλο κλειδί. Παρότι ανησυχώ βαθύτατα σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών και το αν θα γίνουν σεβαστά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης για τη δικαιοσύνη των εκλογών λόγω της καταστολής ε, από πλευρά της κυβέρνησης ε, και που οδηγεί σε περιορισμό της πολυφωνίας και των ανεξαρτήτων μέσων κοινωνική ενημέρωσης στον κόσμο είναι στη δεύτερη τάξη σε σχέση με τους εξορισμένου δημοσιογράφου και τις φυλακίσεις αντιφρονούντων η Αιθιοπία και δεν μπόρεσαν καν να μετάσχουν στην προεκλογική εκστρατεία. επίση ελέγχουν ελέγχεται η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να μην γίνονται συγκεντρώσεις από την αντιπολίτευση και η αστυνομία επίσης ε, έχει ε, διαλύσει ε, φιλινικές διαδηλώσεις σε βασικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαράδεκτες και οφείλουμε να τις καταγγείλουμε επίσημα. Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα θερμά σας λόγια. Ίσως να μην κοιτάω αν έχει περάσει ο χρόνος σας όταν μιλάτε. Και τώρα ο κύριος Επίτροπος. Ο κύριος Επίτροπος Τηγιαννής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση που γίνεται την πιο κατάλληλη στιγμή. Συμφωνώ με τις περισσότερες από τις ανησυχίες που εγείρατε για την εταιρική μας σχέση αλλά αυτή η εταιρική σχέση έχει πολλές πλευρές. Ορισμένες είναι πιο συζητήσιμες από άλλες. Θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη ότι έχουν υπάρξει ουσιώδεις θετικές εξελίξεις για τη χώρα και για το λαό της και τον επικοδομητικό και κρίσιμο ρόλο της στην περιοχή και ευρύτερα. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με την Αιθιοπία και να τονίσουμε ακόμη περισσότερο ότι επιδιώκουμε τον εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών. Όταν ε, θα περάσει ο προεκλογικός πυρετός, θα δεσμευτούμε ακόμη περισσότερο με τις αρχές της χώρας για την μακροπρόθεσμη προσπάθεια εκδημοκρατισμού της χώρας. Εάν η Αιθιοπία θέλει να διατηρήσει τη σταθερότητά της και να επιτύχει το επίπεδο χώρας μεσαίου εισοδήματος μέχρι το 2025 είναι ε, απαραίτητο ο πληθυσμός να έχει δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του. Η Φεντερίκα Μογκερίνη, η εκπρόσωπος, προτίθεται να επισκεφθεί την Αιθιοπία στο εγγύς μέλλον για να διαπιστώσει επιτόπου η ίδια την κατάσταση και να συζητήσει τα θέματα που προκαλούν ανησυχίες σε εμά με τους ηγέτες της χώρας. Σας ευχαριστώ, πολύ, για την προσοχή σας και για αυτή την πλούσια, τόσο πλούσια συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε.